Der Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Τα συνοπτικά πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν έχουν διανεμηθεί. Έχετε παρατηρήσεις, αντιρρήσεις, όχι. Εγκρίνονται λοιπόν τα συνοπτικά πρακτικά.